σημείο είναι η έκθεση Γκαρσές Ραμών, ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για το θεματολόγιο του Ευρωπαίου Καταναλωτή στις 22 Μαΐου του 2012. Η Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ε, Εσωτερική Αγορά και Προστασία του Καταναλωτή ενέκρινε σχεδόν με ομοφωνία ε, την γνώμη τη στι 14 Μαου του 2013. Θέλω να ευχαριστήσω του, τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών και του προσωπικού που συνεισέφεραν έτσι ώστε σήμερα να φτάσει εδώ ένα κείμενο το οποίο θα δώσει πιο ισχυρή φωνή στους καταναλωτές και στις ενώσεις τους για την περίοδο 2014-2020. Οι τρεις βασικοί στόχοι είναι οι εξής. Πρώτον, να ενισχύσουμε την ασφάλεια του καταναλωτή. Δεύτερον, να βελτιωθεί η γνώση του καταναλωτή. Τρίτον, να αυξηθεί η συμμόρφωση και να δοθούν δυνατότητες προσφυγής. Τέταρτον, ε, να βελτιωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να προσαρμοστούν στις κοινωνικές και τις οικονομικές αλλαγές. Η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι βασικές θεμελιώδες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ασκούνται εύκολα και αποτελεσματικά σε βασικούς τομείς όπως ε, η διατροφή, η υγεία, η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές ε, και ψηφιακές υπηρεσίες, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων επίσης είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η καλή ενημέρωση και κατάρτιση των καταναλωτών μειώνει τους κινδύνους εναντί ε, επικίνδυνων ή παραποιημένων προϊόντων καθώς επίσης και έναντι ε, παραπλανητικής διαφήμισης ή κινδύνου από χρηματοοικονομικά προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο η εκπαίδευση θα πρέπει να διαρκήσει όλη τη ζωή των πολιτών και να ξεκινάει από το σχολείο. Η πρόσφατη ε, χρηματοπιστωτική κρίση ε, δείχνει ότι πρέπει οι κατανοητές να ενημερώνονται για τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θα πρέπει οι πληροφορίες που τους δίνονται να είναι πιο αντικειμενικές, αμερόληπτες και να έχουν οι πολίτες περισσότερη πρόσβαση στα μέσα που χρειάζονται για την μια επαρκή επανόρθωση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιωθεί ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών παντού με μέτρα οικονομικά και νομικά μέτρα που είναι απαραίτητα γι' αυτό. Θα ε, πρέπει να τους δίνεται ευκαιρία να συνεργάζονται με τις ε, κρατικές αρχές και να καταγραφούν όλες οι ενώσεις κανονιτών σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κατάλογο. Ε, Επίσης, ε, η ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά ε, θα πρέπει να δίνει στους καταναλωτές ε, να εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους. Σε γενικό επίπεδο οι ευρωπαίοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν καινούριες προκλήσεις όπως για παράδειγμα η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η χρηματοοικονομική απορρίθμιση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η γύραση του πληθυσμού. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει μέτρα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενό ε, μηχανισμού συλλογική αποκατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται περισσότερο αντικειμενικέ, προσβάσιμε και αξιόπιστε πληροφορίε για του καταναλωτέ. Δεδομένου ότι αυξάνονται οι ανισότητε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο την αλληλεγγύη που είναι βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ε, τα στεγαστικά δάνεια και οι αντίστοιχε συμβάσει θα πρέπει να αέρονται όταν υπάρχουν συνθήκες όπως για παράδειγμα ενεργεία που δεν οφείλονται τους ε, καταναλωτές. Ε, θα πρέπει ε, να μπορεί ο καταναλωτής να εξοφλήσει το χρέος του επιστρέφοντας το ακίνητο ή να ρυθμίσει με τρόπο πιο προσαρμοσμένο το χρέος του. Θα πρέπει επίσης ε, να προσέξουμε πολύ τη σήμανση των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό να δίδουμε, να βελτιώσουμε ε, επίσης την ε, ε, κατάσταση των ευάλωτων ομάδων όπως παιδιά, βρέφη, ανάπηροι κλπ. Θα πρέπει να μπορούν ιδιαίτερα αυτοί να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να κινηθούμε έναντι παράνομων πρακτικών που ε, καθιστούν τους ε, καταναλωτές ε, ομοίρους συγκεκριμένων προϊόντων. Στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική καταναλωτή θα, την, θα πάρει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως στη διαδικασία Catch the Πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς ομιλητές και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Σας παρακαλώ να είστε ε, πολύ ακριβείς στο χρόνο σας. Θα είμαι πολύ αυστηρός. Πρώτος ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο εισηγητής. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ε, θέματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη ε, εκ μέρους των πολιτών χώρες ε, όπως η δική μου και άλλες χώρες που περνάνε οικονομική ύφεση ε, είναι χώρες όπου πρέπει να εμφανιστεί η ε, κατανάλωση. Κάποιοι ε, δεν έχουν χρήματα και άλλοι που έχουν δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς ώστε να ξοδέψουν. Ε, γι' αυτό ε, το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης είναι πολύ σημαντικό, ιδίω όσον αφορά την, τις διαδικτυακές τις αναλλαγές. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων φοβούνται να αγοράσουν κάτι από το διαδικτύο γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι οι αγορές αυτές θα είναι ασφαλείς. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να εξασφαλιστεί απαραίτητη προστασία και χαιρόμαστε που αυτό ε, εισάγεται τώρα στο σύστημα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν και την εμπιστοσύνη και τις γνώσεις που απαιτούνται. Επίσης, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι θέμα που αφορά όλη τη διάρκεια της ζωής του καταναλωτή. είναι η διαβίου μάθηση. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε για το χρόνο σα, Ο Κορέα Ντεκάμπο είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκαρσέ για αυτή την έκθεση γνωρίζουμε τα κλασικά παραδοσιακά θέματα προστασίας του καταναλωτή, πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ασφαλείς εμπορικές ε, πράξεις, τα προϊόντα να είναι αξιόπιστα, ασφαλή επίσης. Σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων όμως έχουμε και καινούριες προκλήσεις, καινούρια προβλήματα. Η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση ε, απαιτεί ε, επίγοντα μέτρα προστασίας έναντι χρηματοπιστωτικών ε, ε, πρακτικών που οδηγούν, καθιστούν πιο ευάλωτους ακόμα τους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια στα χρηματοπιστωτικά μέτρα και μέσα και υπηρεσίες. Ε, υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι η βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να προστατεύονται ο κατανοητής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αυτό αποτελεί πρόσθετη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Next speaker is Madame Miranda. Κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Βιθέντε Γκαρσές για αυτή την έκθεση που είναι πολύ επικαιρή. Κέρια στην Ισπανία έχουμε χιλιάδες άτομα τα οποία επηρεάζονται από στεγαστικά δάνεια και την αδυναμία να επιστρέψουν το κινητό τους προς εξόφληση του χρέους. Επίσης έχουμε πολλούς ε, ε, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ε, των οποίων είναι όμοιροι. Ε, έγινε κατάχρηση από πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων της χρήσης και της πώλησης τέτοιων προϊόντων ε, κάποιων προτιμησιακών ε, συμμετοχών σε επιχειρήσεις ε, σε, σε, σε, τα οποία απολύθηκαν σε ανθρώπου, οι οποίοι δεν ήξεραν καλά-καλά να διαβάσουν τη σύμβαση την οποία επέγραφαν. Πολλοί νέου, παιδιά, ακόμα και γέρους θα τους υποστηρίξουμε με τον ταπεινό τρόπο που γνωρίζουμε. Κύριος Φερέιρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ συχνά ε, κάνουμε την υπόθεση ότι όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε την ενέα αγορά, ε, όσο πιο πολύ φιλελευθερωποιούμε την Ευρώπη, όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε τον ανταγωνισμό, τόσο πιο πολύ προστατεύουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή. Λάθος. Μεγάλο λάθος το, δείχνει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι φιλελευθερωποιήσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις βλάπτουν τον καταναλωτή. Ενέργεια, μεταφορές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης η απελευθέρωση των γεωργικών και εμπορικών πολιτικών με διαδοχικά σκάνδαλα ε, και με προβλήματα στην δημόσια υγεία και στην ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει να διορθώσουμε τις βάσεις στις οποίες βασίζεται αυτή η συζήτηση. Αν θέλουμε μια πραγματική προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και όχι αυτά να είναι απλώς η βιτρίνα για τις άλλες μας πολιτικές. Ευχαριστώ. Κυρία Σενιάλοβα. Μια ισορροπημένη πολιτική καταναλωτών στην Ευρώπη θα πρέπει να φροντίζει να δίνει προτεραιότητες ε, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, χρειάζεται καλή λειτουργία του συστήματος με ενημέρωση, δημόσια ενημέρωση των καταναλωτών και των ενώσεων καταναλωτών σχετικά με τα διάφορα προϊόντα θα πρέπει ε, ε, η Επιτροπή να ασχοληθεί με τη διακριτική μεταχείριση που ε, ενίοτε ισχύει έναντι ορισμένων καταναλωτών. Πολύ συχνά υπάρχουν επιθετικές τεχνικές για να επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών, ιδιαίτερα περισσότερο ηλικιωμένων καταναλωτών που είναι περισσότερο ευάλωτη. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο, τον εισηγητή, για την θαυμάσια εισήγησή του. Ευχαριστώ. Κυρία Μπέτζ. Κύριε Πρόεδρε, οι ε, καταναλωτές στην Ευρώπη ε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και λόγω της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμυνθούμε κατά των ε, αθέμητων πρακτικών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τις ε, ενώσεις καταναλωτών. Η έκθεση αυτή φροντίζει να ενημερώνονται κατάλληλα οι καταναλωτές. Εγώ είμαι σύμφωνη με τις προτάσεις του εισηγητού. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα ευρωπαϊκό μητρό και υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητού. Κυρίως θα πρέπει να έχουμε κατά νου την κατασπατάληση τροφίμων. 90 εκατομμύρια τόνοι ε, καταστρέφονται και αυτή η κατασπατάληση δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι καθήκον μας εδώ να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρέντεγκάστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητού Βισέντε Μιγγέλ Γκασές Ραμών σχετικά με την πρόταση αυτή. Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν όλο και περισσότερο να έχουμε κατά νου τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τα δικαιώματα των καταναλωτών διαφορετικά δεν θα είχαν νόημα για αυτούς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο στα πλαίσια μιας άνησης μεταχείρισης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τις πρακτικές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως έναν των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν ε, ε, οικονομικές δυσκολίες και πίεση λόγω ενυπόθηκων δανείων. Είναι τεράστιο το κόστος το οποίο φέρουν οι φορολογούμενοι και ε, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε το να πλήττονται ακόμη περισσότερο οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω καταστάσεων πέραν του ελέγχου τους. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κ. Μπάνγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τα συμφέροντα των καταναλωτών και κυρίως να μιλήσω για τα δικαιώματα των παιδιών, για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να φροντίσουμε στην Ευρώπη να έχουμε κάτι σαν αυτό που έχει η Ελβετία, παραδείγματο χάρη. Ήδη για τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να ε, γίνονται στόχος διαφημίσεων. Δεν θα πρέπει να απευθύνονται διαφημίσεις σε κοινό παιδιών κάτω των 12 ετών. Ε, θα πρέπει και εμείς λοιπόν να σκεφτούμε κάτι αντίστοιχο για να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από προϊόντα καπνού, από υνοπνευματόδη ποτά, ε, προϊόντα που είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Όπως επίσης τα παιδιά θα πρέπει επίσης να καταναλώνουν λιγότερη ζάχαρη και σαχαρόδη προϊόντα. Η κυρία Μπέρες. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al ponente, el señor Garcés. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την πλήρη και ιδιαίτερα αναγκαία έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ατζέντα αυτή την οποία παρουσίασε ο εισηγητή όσον αφορά του καταναλωτέ, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ σημαντικέ προκλήσει, όπω την παγκοσμιοποίηση, τον νέο ψηφιακό χαρακτήρα των οικονομιών μα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε πάρα πολύ γρήγορα να ανταποκριθούμε στι νέε αυτέ προκλήσει. Προσβλέπω λοιπόν στην επόμενη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Από τότε που δημιουργήσαμε την εσωτερική αγορά, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά έχει προχωρήσει πολύ γρηγορότερα από την νομοθεσία εκείνη η οποία προστατεύει και εγγυάται τελικά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προσαρμοστούμε στους νέους καιρούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πιο βιώσιμες μορφές κατανάλωσης στα πλαίσια των οποίων θα προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίω τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων καταναλωτών. Θα ήθελα να δώσω στον Επίτροπο σε τώρα το λόγο για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά την ατζέντα ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Υπάρχουν ε, κάποιες προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας. Και φυσικά υπάρχουν ε, οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεις των οποίων τα σημεία και τις προτεραιότητες έχουμε λάβει υπόψη. Θέλω πραγματικά εδώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ραμόν, καθώς και τους σκιώδες εισηγητές για την εργασία τους. Πρόκειται για πάρα πολύ χρήσιμη εργασία η οποία θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή σαν ε, κατευθυντήρια γραμμή για την ε, από εδώ και πέρα εργασία μας. Ευχαριστώ επίσης και το Συμβούλιο για τον Οκτώβριο θέτησε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, κάτι που πραγματικά συμβαδίζει με την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να λάβουμε υπόψη μας τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές κινητοποιούν την αγορά, η αγορά κινητοποιεί την οικονομία. Και βεβαίως εδώ μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας των καταναλωτών, η ενημέρωση, η εκπαίδευση των καταναλωτών, η στήριξη στις οργανώσεις των καταναλωτών και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία κλειδιά για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και την πολιτική ανατομέα και την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. Ιδιαίτερα λοιπόν θα ήθελα εδώ να εντοπίσω ότι οι υπηρεσίες αυτές οι ψηφιακές, η ενέργεια, οι μεταφορές, καθώς και οι οικονομικές υπηρεσίες που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν προτεραιότητες, καθώς και η προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων καταναλωτών, είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στο επίκεντρο της ε, προσπάθειάς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική για τους καταναλωτές να είναι προς και προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών σε μία περίοδο που πολλοί από αυτούς τους Ευρωπαίους καταναλωτές περνούν δύσκολους καιρούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολίτες μας γνωρίζουν και ε, δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά μέσω της ε, οικονομίας και της ε, καταναλωτική τους δραστηριότητα. Το 2014 θα γίνει η πρώτη έκθεση όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την εξαιρετική έκθεση, η οποία πραγματικά θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην περαιτέρω εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις τελικές σας παρατηρήσεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση από το Συμβούλιο. Μου ήρθε η